Τα πρακτικά και τη συνεδρίαση τη 26η και 27η, καθώ και τα πρακτικά τη εκτατη της συνεδρίαση 25η Ιουνίου και στι 28η Ιουνίου, συγγνώμη, έχουν διανεμηθεί. Ε, sì. Una mozione d'ordine perché ένα διαδικαστικό ζήτημα, διότι όπως υπενθυμίσατε, οι φρικτές επιθέσεις ε, τις οποίες ε, βιώσαμε και ως Ιταλίδα θα ήθελα να ε, αποτίσω φορό τιμής και στους Ιταλούς θύματα του Μπαγκλαντές. Ε, θέλαμε να ζητήσουμε αλλαγή στα κατεπήγοντα, αλλά επειδή δεν προλαβαίνουμε κοινωνικά όρια, ας ε, αποσύρουμε το αίτημά μας και ας θεωρήσουμε ότι αυτό ε, το λεπτό υγιής αποτελεί φόρο τιμής σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή. Ως Ιταλίδα επαναλαμβάνω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των Ιταλών θυμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκαρτίνη που αναφέρθηκε αναφέρετε στα θύματα από τη δική σας χώρα και ασφαλώς αναφερθήκατε όχι μόνο εξ ονόματος των Ιταλών συναδέλφων αλλά εξ ονόματος όλων ημών ότι θα πρέπει να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια προς τα, τους οικείους των θυμάτων από αυτές τις χώρες. Οι αρμόδιες πολωνικές και πορτογαλικές αρχές με ενημέρωσαν για την επιλογή της κυρίας Ούρσουλα Κρούπα και του κυρίου Μανουέλ Αντώνιο Ντοσάντος ε, της κυρίας Κρούπα ε, θα τεθεί σε ισχύ τις 24 Ιουνίου του 2016 θα αντικαταστήσει τον κύριο Βολτσισόφσκι ενώ ο κύριος Ντοσάντος θα αντικαταστήσει την κυρία Φερέιρα και θα τεθεί σε ισχύ από τις 28 Ιουλίου του 2016. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους και να επενθυμίσω ότι θα συμμετάσχουν στο